Άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών. Επιτέλους. Καταρχάν, έγκριση της σημερινής διάταξης, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνεται. του Προέδρου. Περαμένα με τον συγκεκριτή κύριο Βιώτη. Α, ο οποίος ήρθε. Ανακοινώσει για τι αποφάσει των συντονιστών τη 29η Αυγούστου. Τις έχετε στα εγγραφά σας. Αν δεν ε, υποβληθούν αντιρρήσεις, θα θεωρηθεί ότι είναι κρίθησαν. Λοιπόν, επί της ουσίας. Γενικός προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ρούμπιχ ζήτησε να μιλήσει πρώτος, γιατί πρέπει να φύγει σε 10-15 λεπτά και να του δώσω το λόγο για τις, ε, τα άλλα τμήματα του προβλήσμου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, χθε συζητήσαμε με το Συμβούλιο στην Ολομέλεια. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική ούτω ώστε να εξακολουθήσει να είναι σε θέση να λειτουργεί η Κομισιόν και για τα άλλα τμήματα για τα οποία είμαι αρμόδιος. Γενικός μας στόχος είναι να αποκαταστήσουμε τις περικοπές του Συμβουλίου. για να δημιουργηθεί μια βάση διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο για να καταλήξουμε πραγματικά στους αριθμούς. οι γραμμές που δεν ε, αποκαταστάθηκαν από τις ομάδες και τις επιτροπές αποκαταστάθηκαν από εμένα ως εισηγητή. Για τον ε, υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων δέχτηκα μία μείωση γιατί η αύξηση που προβλέπετο ήταν 16 ε, 100, υπερβολική αύξηση και είναι συμβολική αυτή η περικοπή 100.000 μόνο για να δείξω ότι όταν προτείνονται δυσανάλογες αυξήσεις τότε κατά τις διαπραγματεύσεις θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα άρα δεχόμαστε κάποιες περικοπές. Η συμφωνία κυρίων με το Συμβουλίο ισχύει δεν ε, υποβάλαμε τροπολογίες για το Συμβούλιο, για το δικαστήριο. Το πρόβλημά μας είναι ότι λόγω της ε, διαδικασίας Brexit θα έχει πολλή δουλειά το δικαστήριο γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που συνδέονται με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας για τα οποία είναι αρμόδιο το δικαστήριο. Γι' αυτό δεχόμαστε τις ε, τροπολογίες που προτείνει η Τζούρι πάνω και από το σχέδιο του προβλησμού της Επιτροπής με βάση το, στο σημείο 200 και επίσης και για το λογισμικό συνολικά 3 εκατομμύρια πάνω από το σχέδιο προπολογισμού της Επιτροπής και 16 νέες θέσεις. 16 λοιπόν θέσεις επιπλέον και 3 εκατομμύρια. Για το ελεγκτικό συνέδριο επαναφέρουμε την περικοπή, του, δηλαδή ακυρώνουμε την περικοπή του Συμβουλίου για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξίσου και στηρίζουμε και κάποιες εδώ αυξήσεις και πέρα από το, προσχέδιο, το σχέδιο προπολογισμού της Κομισιόν που υπευλήθησαν από άλλες πολιτικές ομάδες 490.000 ευρώ πάνω από την πρόταση της Κομισιόν Περιφέρειες, Επιτροπή Περιφερειών. Ακυρώνουμε την περικοπή του Συμβουλίου και στηρίζουμε την πρόταση των σοσιαλιστών και άλλων πολιτικών ομάδων για μια αύξηση 773.000 πάνω από την πρόταση του Συμβουλίου. Για τον διαμεσολαβητή δεν πρότεινε περικοπή το Συμβούλιο, τα αφήνουμε ως έχει. Ε, επόπτης προσωπικών δεδομένων, είπα, δεχόμεθα την περικοπή 100.000 ευρώ. Δεν στηρίζουμε τις τροπολογίες για ακύρωση αυτής της περικοπής. Για την εξωτερική υπηρεσία, Στηρίζουμε όλες τις τροπολογίες ΑΦΕΤ, απόλυτα. Όπως είπα, ακυρώνουμε και εδώ τις περικοπές του Συμβουλίου και προτείνουμε και πέντε νέες θέσεις. Δύο εκατομμύρια προτείνει η ΑΦΕΤ άνω από το σχέδιο της Κομισιόν. Νομίζω ότι είναι καλή η διαπραγματευτική βάση με το Συμβούλιο. Για το Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι χρειάζονται κάποιες ε, τεχνικές προσαρμογές που είναι δημοσιονομικά ουδέτερες. Και επίσης κάνουμε και κάποιες ε, αλλαγές, δηλαδή καταργούμε την παροχή ύδατος και το πλαστικό. Μετά έχουμε κάποιες τεχνικές προσαρμογές του οργανογράμματος μπορώ να σε ενημερώσω ότι κάνουμε 5% περικοπές στο οργανόγραμμα και στον τομέα των βοηθών και, και στον τομέα των υπαλλήλων και μας επιβεβαίωσε το λεκτικό συνέδριο ότι επιβεβαίωσε ακριβώς τις περικοπές, αλλά θα δούμε αν θα το αμφισβητήσει το Συμβούλιο. Και θα δούμε και την ονομασία ορισμένων γραμμών του προπολογισμού. Μετά οι πολιτικές ομάδες ζήτησαν κάποιες τεχνικές αλλαγές. Οι πολιτικές ομάδες. Έχουμε μια τροπολογία της, ε, του Άλντε για 3,5 άνω του σχεδίου της Κομισιόν Επαναρχόμαστε δηλαδή στην κατάσταση προβλέψεων και τα ποσά που προέβλεπε. Γίνονται κάποιες περικοπές που δεν πρέπει να γίνουν και στηρίζω αυτή την πρόταση. Επίσης, οι ομάδες πρότειναν 46 θέσεις ε, ΑΕΣΤΕ να γίνουν ΑΝΤΕ. Στηρίζω αυτή την πρόταση, είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Επίσης, θέλουν να επαναφερθούν 32 θέσεις οι οποίες είχαν πάει από, την, ε, από τις ομάδες στην διοίκηση μέσω της Πασαρέλας. Τώρα οι ομάδες θέλουν να ε, επανέλθουν από τις αρχές του 19 αυτές οι θέσεις της ομάδες με βάση τη διαδικασία του άρθρου 50. Νομίζω οι θέσεις αυτές προσπαθούν να ε, αντιμετωπίσουν κάποιες αλλαγές στις ανάγκες, ε, Κάποιες θέσεις ε, πηγαίνουν προς τις πολιτικές ομάδες, κάποιες θέσεις πηγαίνουν προς τη δίκηση. Δεν είναι εύκολο για έναν να καταλάβει πώς ακριβώς θα εξισορροπηθούν τα συμφέροντα και των δύο. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να δούμε μήπως θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε μέσω χρήσης του επιδόματος γραμματείας κάποιες δυνατότητες ε, για την ε, πρόσληψη περισσότερων συνεργατών Γι' αυτό το λόγο είμαι σχετικά περιοριστικός. Θα πρέπει να επιτρέψουμε να πληρώνονται σωστά οι συνεργάτες μας, γιατί αλλιώς δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρουμπίχη. Και λοιπόν. τώρα να ακούσουμε τους σκιώδεις για τα υπόλοιπα κεφαλαία να σας παρακαλέσω να επικεντρωθείτε όμως στα δικά σας ε, λόγω του χρόνου. Η κυρία Γκαρτία Θαμπάλ. Ευχαριστώ όταν λέτε τα άλλα κεφάλαια είναι και το κοινοβούλιο. Ωραία. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ο κύριος Ρούμπιχ τα εξέτασε, τα εξήγησε όλα. Και ε, η άποψή μου λήφθηκε υπόψη η άποψη της ομάδας μου. Σε μεγάλο βαθμό έχουμε τρεις μικρές διαφορές. Μία έχει να κάνει με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Υποβάλαμε τροπολογίες που πηγαίνουν παραπέρα από αυτές που δέχθηκε ο εισηγητής. Άλλοι για το διαμεσολαβητή. Στηρίζουμε το αίτημα του Ombudsman να εγκριθούν άλλες δύο θέσεις, γιατί έχει πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Και συμφωνούμε για την περικοπή, για την προστασία των δεδομένων. Συγγνώμη, δεν συμφωνούμε. Τα χρειάζονται αυτά τα λεφτά. Και για το Κοινοβούλιο έχουμε υποβάλει δύο τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική παρενόχληση. Το Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει μια δουλειά για να έχει περισσότερες δυνατότητες και προσωπικό για να καταπολεμήσει την ε, σεξουαλική παρενόχληση αλλά θεωρούμε ότι χρειάζονται περισσότερα. Γι' αυτό υποβάλαμε δύο τροπολογίες που θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες και ελπίζουμε κατά την ψηφοφορία να μας στηρίξουν και άλλες πολιτικές ομάδες. Ο κ. Κόλμελ από το ΕΣΥΑΡΑ. Σα ευχαριστώ πολύ, πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να είμαι σύντομο. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον συνεισηγητή, του συνεισηγητές μάλλον, για την ε, δουλειά που έκαναν, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Εμείς ως SCR ε, συμφωνούμε, μάλλον έχουμε διαφορετικές αρχές. Επί της αρχής διαφωνούμε. Αυτό δεν θα σας εκπλήξει και ανάλογα θα κινηθούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ο κύριο Άλλη από την Άλτε, Δεν ξέρω μήπως θέλει να πάρει το λόγο ο κύριο Τόρβαλτσα. Ε, Δεν γνωρίζω την άποψή του. Ο κύριο Ομάζε από την ΚΟΥΑ. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα κι εγώ. Προσπογράφουμε στις απόψεις του συγητή. Μπράβο του για τη δουλειά του. Γι' αυτό και δεν θα υποβάλουμε τροπολογίες για, τις, για τα υπόλοιπα τμήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους, ο κύριος Τάραντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με την προσέγγιση του συγητή και του κυρίου Ρούμπιχ ιδίω για την ΕΕΔ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Ελληνικό Συνέδριο και το καθεξής. Αλλά ως συνήθως πρέπει να διαχωρίσω τη θέση μου από τη θέση της ομάδας μου. Θέλω να τονίσω την αδιάκοπη, αδιάκοπη ε, και ασταμάτητη και συνεχή στήριξή μου στον καλύτερη χρηματοδότηση των ομάδων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βάλλη από την FTT. Ευχαριστώ. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της συμφωνίας των υπολείπων πολιτικών ομάδων. Έχουμε υποβάλει πολλές τροπολογίες εκ μέρους των συναδέλφων και μου του ιδίου. Για τις δαπάνες νομίζουμε ότι για ορισμένα λύματα είναι απαραδεκτή η αύξηση όπου είχαμε προτείνει 300 εκατομμύρια ε, περικοπές τουλάχιστον για, τα διοικητικές, για τις διοικητικές δαπάνες τουλάχιστον. Εμείς λοιπόν για αυτό το λίμα προτείνουμε μειώσεις εκεί που υπάρχει διασπάθηση και σπατάλη. Και όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα που ζητούν αυξήσει για μα θα πρέπει να κάνουν καλύτερη και χρηστότερη εσωτερική διαχείριση των οικονομικών του και όχι να τα φορτώνουν στου πολίτε που αυτή τη στιγμή κάνουν τόσε θυσίε. διότι δεν δικαιολογείται να ζητάνε αυξήσει στα θεσμικά όργανα όταν σπαταλάνε τόσα ποσά. Δημοσίω ε, θα υποβάλουμε τι τροπολογία από τη φάση. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να έχουμε στηρίξει και από αλλού για να περάσουν και σε ψηφοφορία. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Βάλλη. Ο κύριο Ζάνι δεν φαίνεται να είναι εδώ. Δεν είναι εδώ η αυτή. Είναι και 29 και μπορείτε να φύγετε όπως προβλέπατε στις 9.30 κύριε Ρούμπιχ. Προχωρούμε λοιπόν, δηλαδή πάμε πίσω στην αρχή του προγράμματος, Γενικός Εισηγητής για τον Προπολογισμό του 2019, ο κύριος Βιώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου αμέσως για να μην το ξεχάσω μετά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ρούμπιχ και Γκάγερ. Τον συνάδελφο Γκάγερ που με, με βοηθάνε πολύ για τα υπόλοιπα τμήματα, για τους οργανισμούς και το πώς θα συνθέσουμε την πρόταση για το σχέδιο προπολογισμού του 2019. Η φάση στην οποία βρισκόμαστε και η συζήτηση που έχουμε με τους κοιόδες εισηγητές θα επικεντρωθεί. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και προσπαθούμε να έχουμε μια ερμηνεία του, του από την πλευρά του Κοινοβουλίου που να ακολουθεί τις αρχές και τις προτεραιότητες που είχαμε καθορίσει με την ψηφοφορία του Ιουλίου. Δυστυχώς όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο από την πλευρά του έκανε την πρόταση που όλοι είδατε, χθες την παρουσίασε ο Αυστριακός υπουργό έκανε μια πρόταση που εγώ θα την έλεγα πρόκληση. Χθες το είπα και στην Ολομέλεια στον Υπουργό. Διότι υπέβαλε τον προπολογισμό μιλώντα μόνο για αυξήσει. Αυξήσαμε το ένα, αυξήσαμε το άλλο, είχαμε αυξήσει όλε τι γραμμέ. Προφανώ έκανε σύγκριση με τον προπολογισμό το 18 και το είπα πολύ ξεκάθαρα ότι Έχουμε γυαλιά και βλέπουμε τον προπολογισμό. Προφανώ βλέπουμε με διαφορετική οπτική γωνία τα ποσά του προπολογισμού λοιπόν εμεί. Και βλέπουμε τον προπολογισμό του 19 με γνώμονα και σύγκριση την πρόταση του επιτροπή. Επιτροπής. Είναι πολύ κοινική η προσέγγιση του Συμβουλίου. Τα βλέπουν μόνο από την πλευρά τη, του λογιστική, αυστηρός λογιστική. Χθε λοιπόν ήταν καλή ευκαιρία να έχουμε τον Αυστριακό Υπουργό που το έλεγε για τους πολίτες ουσιαστικά που βλέπω στην τηλεόραση, στο ίντερνετ, στο streaming. Τον άκουγα να λέει τα αυξήσαμε όλα και ο εισηγητής του Κοινοβουλίου έλεγε το αντίθετο, τα περικόψατε όλα θα ήταν αρκετά ευχάριστο για όποιον το άκουγε. Ε, προσπαθήσαμε λοιπόν να εργαστούμε ακολουθώντας κάποιες αρχές. Πρώτα απ' όλα, να επαναφέρουμε τα ποσά που περιέκοψε το Συμβούλιο αδιακρίτως στο σχέδιο προπολογισμού που είχε αρχικά υποβάλει η Επιτροπή. Επίτα ακολούθησε και μια άλλη αρχή. Αρχή που καθόρισε το ίδιο το Κοινοβούλιο και μια αρχή που θεώρησα και εγώ σημαντική. Δηλαδή, πάκτα σερβάντα σουν, ε, θα πρέπει να, να τηρούνται τα συμπεφωνημένα. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν ε, συμφωνήσει ότι θα γίνει με το εργαλείο για την Τουρκία. Τα ποσά λοιπόν πρέπει να πάνε δύο τρίτα από το Συμβούλιο και ένα τρίτο από το κοινοτικό προπολογισμό. Σύμφωνα με την νέα ερμηνεία του Συμβουλίου δεν είναι έτσι. Γι' αυτό εγώ θέλω όσα συμφωνήθηκαν να τηρηθούν. Έτσι καθόρισε και το Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό ακολουθήσαμε τι παλιέ συμφωνίε για να κάνουμε τι προτάσει μα χθε, σε συνεργασία με τον Επιτρόπο που μα βοηθάει πάρα πολύ. Είπαμε, είπε εκείνο δηλαδή, ότι ελπίζω να βρεθεί ένα σημείο σύγκληση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Εγώ επανέλαβα ότι το μόνο σημείο σύγκληση στι θέσει των δύο είναι να τηρηθούν ακριβώ όσα είχαν συμφωνηθεί στο παρελθόν. Αυτά ως προς το... τις αρχές του Κοινοβουλίου. Τώρα για τον προπολογισμό για... υπήρξαν πάρα πολλές προπολογίες και βάσει της αρχικής πρότασης της Επιτροπής που όμως με τους συνεργάτες της με βοήθησε πάρα πολύ για ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς και προσπαθήσαμε ως το δυνατόν να σεβαστούμε αυτό που είχαμε καθορίσει ως στόχο. Φυσικά δεν μπορούμε με το ίδιο πάπλωμα να τα σκεπάσουμε όλα, όπως λέμε στην Ιταλία. Δεν χωράνε όλοι κατά την ίδια κουβέρτα. Αλλά είχαμε και πολλοί επικοδομητικές προτάσεις από μεμονωμένους βουλευτές σε σχέση με τη διόρθωση της πρότασης του Συμβουλίου σε όλες μας τις ε, συνεδριάσεις και τις παρουσιάσεις του προπολογισμού την περασμένη άνοιξη σε διάφορες επιτροπές. Ακούσαμε πώς τοποθετήθηκαν οι διάφορες πολιτικές ομάδες. προσπαθώντας να συνδυάσουμε και να συμπαρασύρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές και πολιτικές ομάδες. Εδώ λοιπόν μερικά παραδείγματα για το Εράσμους υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα αιτήματα από συναδέλφους. Από την Άλντε, από τη δική μου την πολιτική ομάδα ή ξέρω εγώ αυτό που ζήτησε η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Θελήσαμε να υπάρχει αύξηση 15% για το Εράσμος στην πρόταση προπολογισμού μας. Είναι σημαντικό αυτό. Σοβαρή αντίγραφη. Και όπως για τις γραμμές που περικόπτονται από λόγο του εύση, κοιτάζουμε να υπάρξει κάλυψη της διαφοράς. Ακόμη και στο επίπεδο της ε, πρωτοβουλίας για τους νέους και της δουλειάς που θέλει να κάνει το Κοινοβούλιο για την νεολαία μας προτείναμε αύξηση και άλλες πολλές πρωτοβουλίους. Ε, στη γραμμή 2 προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε αιτήματα που μας ήρθαν από τις πολιτικές ομάδες και να καλύψουμε όσα δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην αρχική σύνταξη της πρότασης για το σχέδιο προπολογισμού. Βέβαια, έκανα τι προτάσει μου ανάλογα με το περιθώριο που ήθελα να αφήσω και στην Επιτροπή να αντιδράσει. Γιατί, όπω ξέρετε, τον Οκτώβριο θα έχουμε την ενδεικτική, την, αποστολή, την επιστολή με τι ε, προθέσει που θα μα ε, υποβάλει η Επιτροπή και κάποιου αρχικού και κάποιου νέου υπολογισμού για τα ποσά. Τώρα, για τι προτάσει ε, των φιλελευθέρων για το κοινωνικό ταμείο ή του οργανισμού, δεν θα μπω στι λεπτομέρειε, γιατί το κάνει εδώ ο κύριο Γκάγερ αυτό. Δεν σχολιάζω. Αλλά Απαντήσαμε σε πολλά αιτήματα λόγου χάρη σε αυτά της Επιτροπής Πολιτισμού. Δύο λόγια ακόμα για τη γραμμή 4. Δεν θέλω να μονοπολίσω εγώ τη συζήτηση. Mm. Ε, για τη γραμμή 4 χθες Μπόρεσα να συνομιλήσω με τον ε, Αυστριακό Υπουργό της ε, Εναλλασσόμενης Προεδρίας και ήθελα να σας επισημάνω ότι ο Υπουργό θα παίρνει μέρος στις συζητήσει. Είναι η πρώτη φορά από τότε που συμμετέχω στην Επιτροπή αυτή και παρακολουθώ τα θέματα του προπολογισμού που βλέπω υπουργό τόσο παρόντα και τόσο πρόθυμο να συμμετάσχει στις συζητήσεις. Αυτό μας εξυπηρετεί ε, φοβερά στη συνεννόηση. Δηλαδή και από τεχνικής πλευράς ε, μπορούμε να δώσουμε την κατάλληλη στήριξη στα επιχειρηματά μας και στις λύσεις που βρίσκονται. Οπότε θα βρεθούμε στο δυνατόν πιο συχνά και θα ενημερώνεστε συστηματικά κι εσείς. Χθες τόνισα στον Υπουργό ότι αν έχουμε μια κοινή θεώρηση Κοινοβουλίου κρατών μελών για το τι θέλουμε να γίνει, και ενώ Είπαμε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τα γενεσιουργά αίτια της στόχιας και της μετανάστευσης ε, με τις κλιματικές αλλαγές, τους λοιμούς και ούτω καθεξής. προτεραιότητα της δικής μου κυβέρνησης, της αυστριακής κυβέρνησης και ένα σωρό ε, άλλων κυβερνήσεων είναι αυτό ακριβώ. Αλλά πρέπει τότε να επενδύσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ανθρωπιστική βοήθεια, υποστήριξη το ένα το άλλο χωρίς να προοικοδοτήσουμε όλα αυτά με χρήματα. Αυτό πρέπει να καταλάβει το Συμβούλιο. Ε, αυτήν την γραμμή προσπαθήσαμε να περάσουμε και θέλουμε να αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα ποσά στι διάφορες γραμμές. Για την ανθρώπινη ανάπτυξη, τις εταιρικές σχέσει, την εταιρική σχέση Βορρά-Νότου, την δουλειά που έγινε στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια. Αυτό που επιζητούμε και προσπαθώ να το πω ε, από τη δική μου προσωπική σκοπιά, ε, παρόλο που είναι δική μου πεποίθηση, αυτό που θεωρεί κάποιος εισρωή από από τον έξω κόσμο προς την Ευρώπη μπορεί να προληφθεί στην πηγή του προβλήματος. Αυτό μπορεί να γίνει σε έναν βαθμό με αυτόν τον προπολογισμό, με συγκεκριμένα εργαλεία και μέσα, αλλά πρέπει να γίνει και με συγκεκριμένε επενδύσει από αυτή τη γραμμή. Αυτά είναι όσα ήθελα να σα πω στη γενική παρουσίαση τη δουλειά που κάνουμε και τη πρόταση προπολογισμού που συζητιέται με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Βεβαίως ε, παραμένω στη διάθεσή σας γιατί με ενδιαφέρουν πολύ οι παρεμβάσεις και οι παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Οι σκιώδες ε, από το ΕΛΚ, κυρία Χόλμα, έρχεται το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, καταρχάς, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον συνάδελφο Ντανιέλε Βιώτη για την καλή συνεργασία και να ευχαριστήσω και τους άλλους κοιόδες. Προσπαθούμε να βγούμε από μια δύσκολη κατάσταση. Το Συμβούλιο προσπαθεί να διατηρήσει ένα περιθώριο, ένα περιθώριο λιγμού, όπου όμως δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια. Έχουν εξαντληθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αναπτυξιακής βοήθειας, σε όλους αυτούς τους τομείς όπου υπάρχει σημαντική ανάγκη. Και προφανώς όλοι αυτοί οι τομείς της ασφάλειας ε, πρέπει να υπάρχουν ε, προσαυξήσεις. Πιστεύω ότι μετά από τις χθεσινέ συζητήσει υπάρχει μια ανάγκη να συζητήσουμε λίγο παραπάνω και θέματα εξισορρόπηση του DCI, τη Ευρωπαϊκή ε, Γειτονία, Θα πρέπει να βρούμε καλύτερε ισορροπίε, θεωρώ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να στραφούμε και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μάθουμε τι γίνεται στον Frontex μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί και εγώ προφανώς χθε άκουσα την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης και μέχρι το 2020 αναφέρθηκε 10.000 επιπλέον θέσεις. Μα θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, γρήγορα μάλιστα και τι θα γίνει από δημοσιονομικής άποψης. Τον Οκτώβριο στο διευθυντικό προπολογισμό θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά γιατί το 2020 Πώς θα βρούμε με μιας 10.000 επιπλέον ανθρώπους. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι πολύ απίθανο. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε τον Οκτώβριο, λοιπόν. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει. Γιατί όλα αυτά μας απασχολούν και εμάς και προφανώς θα έχουν να κάνουν και με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να μας πει τι φαντάζεται. Επίση. Ε, έχουμε και μερικέ εξωτερικέ υπηρεσίες, οι οποίες δυστυχώ. παρά το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν οι ανάγκε τους, δεν έχουν αναγνωριστεί. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. από την Ιεμένη, το Ιράκ, το Μπαγκλαντές, ε, τι κονδύλια μπορούν να, να αφαιρεθούν. Γιατί προφανώς και εκεί υπάρχουν κρίσιμες καταστάσεις και δεν είναι μόνο η Βόρειος Αφρική αυτή που πλήττεται και η Αφρική εν γέννη. Άρα να βρούμε μια σωστή ισορροπία. Θεωρώ ότι σε πολλούς άλλους τομείς έχουμε πετύχει το, την κατάλληλη ισορροπία και στην άλλη πιστεύω ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα και σωστά στοιχεία και νομίζω ότι η Ντανιέλα θα κάτσουμε να συζητήσουμε και θα καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Από το ECR, ο κ. Κόλμελ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ σύμφωνο με την ε, προλαλή σα και θα ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Ήταν πολύ εκτενή η δουλειά που έκανε και θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω το εξή. Εδώ μου προκαλεί έκπληξη σχεδόν το γεγονό ότι συμφωνούμε. Και εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δαπανίσουμε πολύ πιο πολλά κονδύλια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη για τον τομέα της μετανάστευσης και μάλιστα για την πρόληψη τη μετανάστευση. μετανάστευσης. Γιατί προφανώς αυτό είναι ο τρόπος να καταφέρουμε οι άνθρωποι αυτοί να μην ξεκινάνε καν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι. Είμαι τεταθειμένος λοιπόν να ταπανίσουμε κονδύλια, αν παράλληλα ως Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήσουμε και νόμιμες ε, οδούς για το άσυλο, για τους ζητούντες άσυλο και τους ε, μετανάστες. Ε. Γιατί στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και ξέρουμε ότι αυτό μας κάνει ευάλωτους. Δεν θέλουμε, δεν τολμάμε να πάρουμε τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε για να βοηθήσουμε του ανθρώπου αυτού. Και εδώ πραγματικά είμαι διατεθειμένο να δαπανίσουμε πολύ πιο πολλά κονδύλια, πολύ παραπάνω από ό,τι σήμερα, αλλά να λειτουργεί το σύστημα, να υπάρχει μια νόμιμη οδός. Όσο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ουσιαστικά εμ, καταπολεμούμε τα συμπτώματα και όχι την αιτία. Και αυτό δεν προτίθεμε να το συνεχίσουμε. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεπρέ είναι σε άλλη συνεδρίαση. Μήπω θα ήθελα να πάρει το λόγο ο κ. Στόρβαλτσα. Ε? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βιώτη για τη δουλειά που έκανε. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Ο κύριος ε, Ντεπρέ είναι, έχει τα πάντα υπό έλεγχο, συνήθω. Αυτό που θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε είναι το εξή ότι θα υποστηρίξουμε τις τροπολογίες μας σε ό,τι αφορά και το τμήμα 1α. Προφανώς ο ορίζοντας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά το mainstreaming για το κλίμα. Και αυτό μας απασχολεί. Θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά και προφανώς ε, σε ό,τι αφορά τη διαμάχη με το Συμβούλιο για το τμήμα 1α, ό,τι μπορεί να κάνει ο εισηγητή να είναι βέβαιο ότι θα τον υποστηρίξουμε. Δεν θα σα ευχαριστήσω στα σβηδικά γιατί μιλήσατε αγγλικά την άλλη φορά. Για την ΚΟΕ δεν βλέπω τον κύριο Νεριάντα. Στου ε, πράσινου έχει φύγει ο κύριο Τάραν. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ανταυτού. Α, συγγνώμη. Uh, Ευχαριστώ. Μας ανησυχούν ε, οι πολύ εκτεταμένες περικοπές στις πιστώσεις υποχρεώσεων που λέει ότι που δεν αιτιολογούνται από το ποσοστό απορρόφησης έτσι οι υποχρεώσεις είναι λιγότερο από 1% του GNI των κρατών μελών με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι το Συμβούλιο θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο Κοινοβούλιο για το επόμενο πολιτές πλαίσιο. Ναι. Καλές όμως είναι οι τροπολογίες ε, του συγητή, οι συμβαστικές. Εμείς ε, υποβάλαμε τροπολογίες ε, για την απασχόληση των νέων, τον έρασμο, το ζωή συν, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανάπτυξη και τη συνεργασία και περαιτέρω στήριξη της Ούνρα και για τα κλιματικά θέματα. Και χαίρομαι που σχεδόν όλες συμπεριλαμβάνονται στις πρώτες αυτές συμβαστικές προτάσεις Ιδιαίτερα μας χαροποιεί η έγκριση για τον πολιτισμό, για τα ανθρωπιστικά, για την ανάπτυξη και κυρίως για τα κλιματικά θέματα. Και θα τα πούμε στις περαιτέρω συζητήσεις των ε, σκιωδών και να δούμε πώς θα πάνε οι περαιτέρω διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σολέ. Ευθυντή παρακαλώ. Ευχαριστώ. Άκουσα με προσοχή την ε, ερμηνεία του εισηγητή. Θα συμφωνήσω σε κάποια σημεία γιατί οι προτεραιότητες που ανήκει, λέει, είναι προτεραιότητες και πολλών κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίως σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές. Ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί κυρίως στα γενεσιουργά του αίτια. Πρέπει λοιπόν να, να αφιερώσουμε κονδύλια για την καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτίων με τρόπο διαφανή και ε, σαφή. Εδώ την θέση αυτή μπορούμε να τη συμμεριστούμε. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένα κονδύλια τα κοινωνικά προβλήματα συγκεκριμένων χωρών, ιδίω των χωρών του Νότου της Μεσογείου, ε, με σοβαρά προβλήματα ανεργίας και προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση εκεί που οι πολιτικές της Ευρωζώνης δεν έχουν ε, φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, υποβάλαμε τροπολογίες για να δώσουμε ένα μήνυμα, διότι οι θεσμοί έπρεπε να οργανωθούν καλύτερα στην εσωτερική τους διαχείριση και τις δαπάνες τους. Ε, στο Κοινοβούλιο εδώ θα έχουμε, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη πρόκληση του Brexit. Θα χάσουμε καμιά πενταριά βουλευτές. Πώς γίνεται να αυξάνονται οι διοικητικές δαπάνες σε αυτή την περίπτωση. Εάν θέλουμε στο λίγο των δαπανών να έχουμε αυξήσεις, θα χάσουμε την εξοπιστία μας και πάνω απ' όλα θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι ενώπιον των πολιτών. Θέλουμε να γίνει κατανοητό ότι οι αυξήσει που ζητάμε σε κάποια λύματα του υπολογισμού ε, δικαιολογούνται και ότι κάνουμε πολύ σωστή εσωτερική διαχείριση στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Για τις προτάσεις λοιπόν του συγγητή ε, σε πολλά συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να είμαστε και πιο πραγματιστές. Ευχαριστούμε και για την ΕΝΕΦ. E δεν νομίζω ότι βλέπω τον κύριο Ζόλτεκ. Ωραία, οπότε ολοκληρώνουμε με τον γύρο των σκιωδών σε ό,τι αφορά άλλα μέλη, ο κύριος Γκάιερ για τους οργανισμούς. Ευχαριστώ, ναι, για τους εξωτερικούς οργανισμούς. Ναι, έτσι δεν είπατε. Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι. Λίγα λόγια για την κατάσταση του προπολογισμού για τους εξωτερικούς ε, οργανισμούς. Είμαι σε επαφή μαζί τους, ώστε να μαθαίνω απευθείας πώς ε, εκτιμά ο κάθε τέτοιος οργανισμός τον προϋπολογισμό σε σχέση με τις ανάγκες του. Δεν θεωρώ. ότι η Κομισιόν ε, ε, έχει λάβει υπόψη αυτά που θεωρούν αναγκαία οι οργανισμοί για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Υπάρχουν έξι συγκεκριμένα φορείς τέτοιοι. που ζήτησαν περισσότερο προσωπικό ή περισσότερες πιστώσεις από αυτά που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού. Εκτός από αυτούς τους έξι φορείς, επανήλθαν, ε, ακυρώθηκαν οι περικοπές για να ληφθεί υπόψη και το αίτημα των ε, φορέων. Και υπάρχουν μία-δύο ειδικέ περιπτώσεις όπου τη στιγμή που δημοσιεύθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού, δεν είχε ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος ο οποίος οδήγησε κατόπιν ο τριμερής διάλογος για κάποια θέματα. Θα ήθελα να σας πω, αλλά δεν θυμάμαι τώρα αμέσω ποιοι είναι αλλά μετά την ολοκλήρωση κάποιων τριμερών διαλόγων οι ε, οργανισμοί αυτοί έχουν επιπλέον αρμοδιότητε που δεν ανακλούνται λοιπόν στο σχέδιο προπολογισμού. Εκεί πρέπει να δούμε συγκεκριμένα πώς θα ενισχύσουμε τους πόρους αυτών των προπολογισμών, των ε, οργανισμών. Αυτό θα προτείνω για το Κοινοβούλιο. Να πω όμω κάτι για την Frontex. Πρόσφατα πήγα στη Βαρσοβία και συζήτησα με την Frontex και είδα τις ανάγκες για το εγγύς μέλλον. Είναι σαφές. Με κάθε συμφωνία του Συμβουλίου για διαχείριση συνόρων αυξάνονται οι υποχρεώσεις της Frontex, άρα χρειάζεται περισσότερο προσωπικό και περισσότερες πιστώσεις. Όταν γίνεται λόγος για 10.000 δεν είναι 10.000 άτομα τα οποία τα έχουμε ε, κάπου ε, χωρέσει στη Βαρσοβία και μόλις θα ζητάει κάποιο κράτος μέλος κάτι θα τους στέλνουμε κάποιους. Κοιτάξτε, η κατάσταση έχει ως εξής. Η Frontex έχει δικαίωμα να ζητήσει από τα κράτη-μέλη υπαλλήλους των εθνικών συνοριοφυλακών, για παράδειγμα της γερμανικής συνοριοφυλακής ή της γερμανικής αστυνομίας, για να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκή επιχείρηση κάπου όπου υπάρχει κρίση. Χρειάζεται πόρους το Frontex ε, σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά δεν θα χρειαστεί να προσλάβει 10.000 άτομα η Frontex. Βεβαίως θα αυξηθεί το προσωπικό, ναι, αλλά δεν θα αυξηθεί κατά 10.000 από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά αυτό που για πρώτη φορά ε, χρειάζεται και δικούς της πόρους. Μέχρι στιγμής έκαναν αναβλώσεις, ε, ενοικιάσεις, αλλά χρειάζονται και ένα μόνιμο εξοπλισμό. Χρειάζεται για παράδειγμα τζιπ, ε, χρειάζεται κάθε είδους ε, εξοπλισμό που μέχρι στιγμής ε, τους, ε, τον διέθεταν ε, τα κράτη-μέλη και πρέπει να παρακαλέσουν και σε ορισμένε περιπτώσει ήταν και ακατάλληλο. Είναι πολύ πιο απλό και πιο οικονομικό να νοικιάσεις ένα ελικόπτερο επιτόπου παρά να ζητήσεις από την Σουηδική συνοριοφυλακή να στο στείλει στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Αλλά δεν υπήρχαν λόγοι για να αγοράσει μέχρι τώρα κάτι τέτοιο η Frontex. Τώρα όμως αλλάζει η κατάσταση. Γι' αυτό υπάρχουν επιπλέον ανάγκες. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ισχύσουν οι τάξεις μεγέθους που αναφέρθησαν. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιες επιτροπές δουλεύουν πολύ στενά, συνεργάζονται πολύ στενά με ορισμένους εξωτερικούς οργανισμούς. Έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες του κάθε, της κάθε επιτροπής. Αλλά δεν είναι δυνατόν η γνωμοδότηση κάθε επιτροπής να ζητάει περισσότερους υπαλλήλου και περισσότερους πόρους από ε, όσους ε, ζητάει και θεωρεί αναγκαίους ο ίδιος ο οργανισμός. Είναι πολύ δύσκολο σε μια διαπραγμάτευση κατόπιν, για παράδειγμα, να λέμε θέλουμε 50 παραπάνω θέσεις για την ΕΑΖΟ και άμα δούμε τι έχει ζητήσει η ίδια η ΕΑΖΟ να δούμε ότι είναι 25. Ε, αυτό αποδυναμώνει τη θέση μας. Καταλαβαίνω ότι ε, το Κοινοβούλιο θέλει να στέλνει ορισμένα μηνύματα. Κάποιοι θεωρούν ότι κάποιος οργανισμός δουλεύει πολύ καλά, άρα πρέπει να τον ενισχύσουμε. Έχω κάποια κατανόηση για τέτοιου τύπου ε, ενέργειες, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην έχετε συνοηθεί προηγουμένω με τους οργανισμούς. Δεν μπορεί να περάσει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό Δεν στηρίζω τα αιτήματα κάποιων ε, επιτροπών για την επέκταση των δραστηριοτήτων κάποιων οργανισμών. Γιατί τη συνέκρινα με τι απαιτήσει των ίδιων των οργανισμών και ήταν υψηλότερε. Άρα δεν μπορώ να τη στηρίξω. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Χόλμαϊ. Συγγνώμη, ε, συνάδελφε Γκάιερ. Υπάρχουν συνάδελφοι Και εμεί και ο συνάδελφο Ντεπρέ είμαστε σε επαφή με του οργανισμού για την Frontex και τον ΕΑΣΟ. Θα ακούσω πρώτα απ' όλα την απάντηση τη Κομισιόν. Τι θα προκύψει τον Οκτώβριο. Δεν έχει έννοια να επιχειρούμε εμεί να καταλήξουμε. Πρέπει να δούμε την πλήρη πρόταση της Κομισιόν. Και για την ΕΑΣΟ, και για τα καθήκοντά της, και για το προσωπικό που χρειάζεται, και για την Frontex. Σίγουρα δεν περιμένουν κάπου 10.000 άτομα στην Βαρσοβία, αλλά κάποιοι είναι ήδη στη Βαρσοβία και έχουν ε, πολλά προβλήματα. Ο κύριος Σιτόρσκι το ξέρει. Δεν έχουν επαρκές προσωπικό. Δεν έχουν δυνατότητα να επικοινωνήσουν τα κράτη-μέλη, να λύσουν κάποια διοικητικά θέματα και χρειάζεται να κάνουν πολλές προσπάθειες και αν ήδη και αν θα πρέπει να αναλάβουν την ε, διοίκηση και επιπλέον 10.000 ατόμων εκ των οποίων κάποιοι θα αποσπαστούν από τα κράτη-μέλη και κάποιοι θα πρέπει να προσληφθούν από τη Frontex την ίδια, αυτό θα σημαίνει τεράστιο διοικητικό άχθος. Αλλά η Κομισιόν θα πρέπει, όπως και για το ΕΑΣΟ, να μας πει εάν θα μας κάνει μια πρόταση για τον ε, Οκτώβριο. Για το Εουλίζα. Στην Γκάιλ, δεν συμφωνώ. Γιατί το συζήτησα αναλυτικά με την Εουλίζα. Και το κύριο πρόβλημά τους είναι ότι πρέπει να κάνουν πολλές προπαρασκευαστικές εργασίες για την EAS ε και ο Τόμας με άκουσε, τους ακούσαμε μαζί και όλες οι πολιτικές ομάδες διαπιστώσαμε τις ανάγκες της ΕΟ Λίζα. Γι' αυτό θα παρακαλούσα να το συζητήσουμε με την ησυχία μας λίγα και αυτό το θέμα. Για τη Frontex και την ΕΑΣΟ θα πρέπει να περιμένουμε τον Οκτώβριο. Για την ΕΟ έχω πολλές αμφιβολίες. Γιατί δεν τα καταφέρουν με τα τόσα καθήκοντα που έχουν. Πρέπει νομίζω με την ησυχία μα να το ξαναδούμε και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλει κανεί άλλο το λόγο, λέει ο πρόεδρο. Δεν βλέπω κάποιον άλλον, αλλά ήθελα και εγώ να συμπεριλάβω τον εαυτό μου στον κατάλογο των απορριτών. Έχω μια-δύο ερωτήσει προ τον κύριο Βιώτη. Πρώτον, για το αποθεματικό για την κρίση, της, για τις ενδεχόμενε κρίσει στη Γεωργία, το γεωργικό τομέα. Δεν βλέπω τίποτε στις συμβιβαστικέ σας προτάσεις γι' αυτό. Και ήθελα απλώ να μου πείτε ποια είναι η συλλογιστική. Και το άλλο είναι τα 25 εκατομμύρια περικοπές στη συνεργασία με τη Μεσανατολή. Ε, αυτή που έγινε από το Συμβούλιο. Φαίνεται να μην το πειράζουμε καν. Ε, για αυτά τα δύο θέματα ήθελα μια διευκρίνηση από sua ναι, αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, Πρόεδρε, με ρωτάτε για το αποθεματικό, ε, για, το, για τη γραμμή 2, για το heading 2, για τη Γεωργία. Εκεί αφήσαμε... Τίτλο. Εδώ τα αφήσαμε τα 200 εκατομμύρια στη γραμμή 2, αν αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, αλλά ο σκοπός ήταν να γίνει αύξηση, να το μεγαλώσουμε το ποσό. Διότι θέλουμε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες κρίσεις που βλέπουμε να υπάρχουν στο γεωργικό τομέα. Ναι, αυτό το ποσό το αφήσαμε, αλλά εάν το ζητάει η Επιτροπή μπορούμε να, την, ε, να το παίρνοντας κονδύλια από άλλες γραμμές. Μπορούμε να αυξήσουμε αυτή τη γραμμή. Αυτή την πρόταση, αλλά θα πρέπει να πάρουμε κονδύλια από άλλες γραμμές. Σε ό,τι αφορά τις περικοπές για τη Μέση Ανατολή, αυτό που ρωτήσατε εσείς, αυτές τις περικοπές τις ζήτησε δική μας Επιτροπή, η Επιτροπή ΝΤΕΒΕ και σκεφτήκαμε να ακολουθήσουμε την γραμμή της, της αρμόδιας για αυτή την πολιτική επιτροπή. Ωραία. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Κάποιος άλλος. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση θα δώσω το λόγο στον κύριο Βιώτη αν θέλει να ανακεφαλαιώσει Mr. Viotti, Θέλετε να συνοψίσετε, κύριε Βιώτη, να πείτε μια τελευταία κουβέντα. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, ζητάει το λόγο και η Επιτροπή για να απαντήσει σε ένα-δυο παρατηρήσεις που έγιναν, οπότε πριν από εσά σας ακούσουμε την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να με συγχωρείτε, κύριε Βιώτη. Αλλά η κυρία Χολμαγέρ έθεσε ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συντομεύω. Πράγματι, οι νομοθετικές προτάσεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή χθε και ανακοινώθηκαν και από τον πρόεδρο Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, θα έχουν επιπτώσεις και στον προπολογισμό το 2019, ναι. ιδίω στην Frontex και την EASO. Θα δούμε πώς θα το συμπεριλάβουμε στην διορθωτική επιστολή του Οκτωβρίου, αλλά δείτε τι ε, κονδύλια διατίθενται ήδη για αυτούς τους οργανισμούς, για να μπορείτε να αποτιμήσετε αν ε, οι προστασιανάκες τους πρέπει να καλυφθούν. Τώρα για την ε, Frontex από τους 10.000 συνοριοφύλακες. Εκτιμούμε ότι η διαδικασία της συναπόφασης για την έγκριση της νέας αυτής πρότασης θα χρειαστεί χρόνο. και εκτιμούμε ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις το 2019 θα είναι σχετικά περιορισμένες, διότι θα αρχίσουν να φαίνονται στο δεύτερο μέρος της χρονιάς κυρίως, στο δεύτερο εξάμεινο. Αυτά που είπε και ο κύριος Γκάγερ, θα υπάρξουν διαφορετικές κατηγορίες ε, μεταξύ αυτών των 10.000 συλλογοφυλάκων και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε όταν συζητηθεί η πρόταση εδώ, στην Επιτροπή σας. Όμως, υπάρχει μια κατηγορία ε, υπαλλήλων που θα χρειαστεί χρόνος να την, ε, για να προσλάβουμε τους απαραίτητους. Μετά θα υπάρξουν αποσπασμένοι συνοριοφύλακες, μια άλλη κατηγορία, εκεί όπου τα κράτη-μέλη θα λάβουν οικονομική αποζημίωση εφόσον ε, χρειαστεί να προσλάβουν αντικαταστάτες για αυτούς τους αποσπασμένους και μετά θα έχουμε και μια τρίτη κατηγορία αποσπασμένους ενεροφύλακες που θα ε, Του καλούμε μόνο σε περίπτωση που υπάρχει πραγματική κρίση. Αλλά αυτά μπορούμε να τα δούμε και σε επόμενο στάδιο. Το μεγαλύτερο δημοσιονομικό αντίκτυπο θα τον αισθανθούμε το 2020 και θα φανεί και στο σχέδιο υπολογισμού του χρόνου, την άνοιξη του χρόνου. Εάν θέλουμε να φτάσουμε τα 10.000 άτομα για τις τρεις κατηγορίες προσωπικού το 2020, θα πρέπει να ανασκουμποθούμε. Το 2020 λοιπόν θα υπάρχει σοβαρότερη ε, ο σοβαρότερο αντίκτυπο. Ευχαριστούμε και τώρα εσεί, κύριε Διώτη. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ τη γραμματεία που με επισήμανε ότι παρεμήνευσα την ερώτησή σας, Πρόεδρε, για το αποθεματικό για τις κρίσεις. Σήμερα δεν γίνεται να υπάρξει, να, υπάρξει αύξηση, διότι βάσει του κανονισμού προβλέπεται ήδη βάσει των όσων ορίζει η ΚΑΠ. Δεν μπορούμε τώρα να, να παρέμβουμε σε επίπεδο σχεδίου προπολογισμού στη δημοσιονομική αυτή γραμμή για να ψηθεί το αποθεματικό για τι κρίσει. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είχα καταλάβει την ερώτησή σα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα γενικά μου συμπεράσματα, πολύ πολύ γρήγορα, ευχαριστώ του ε, σκιώδει συναδέλφου που εκτιμούν γενικώ από ό,τι ακούσαμε τη δουλειά μα. Μα φτάσαν φυσικά στα χέρια μα κάποιε προτάσει, κάποιε τοπολογίε. Ακούσαμε τι προτεραιότητε των διαφορετικών πολιτικών ομάδων, αλλά νομίζω ότι είμαστε στη σωστή οδό για να φτάσουμε σε συμφωνία που θα μπορούσε να του εκφράζει όλου. Τι ερχόμενε ημέρε, τι επόμενε συνεδριάσει μα και συναντήσει Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε και τις μικρές αποκλίσεις στην ερμηνεία κάποιων αριθμών, κάποιων ποσών, κάποιων προτεραιοτήτων που μπορεί να υπάρχουν ακόμα και πάλι ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Βιώτη. Η ψηφοφορία προβλέπεται στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες και στην Ολομέλεια στις 24 Οκτωβρίου εδώ στο Στρασβούργο. Μετά θα ξεκινήσει στις 7 Νοεμβρίου η διαδικασία συνδιαλλαγής. Αυτό ήταν το σημείο 3. Και να περάσουμε στο 4 λοιπόν τώρα. Δημιουργία της διευκόλυνσης ε, για τη διασύνδεση της Ευρώπης. Η κυρία Βάιντερε είναι η συγκήτρια. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πέτρη, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότηση για τι δημοσιονομικέ πτυχέ σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για το Connecting Europe Facility για την περίοδο μετά το 2020. Τα γνωρίζετε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη σχετική προτάση στις 2 Μαΐου του τρέχοντος έτου και προτείνει λοιπόν έναν φάκελο 42,3 δισεκατομμύρια σε τρέχουσες τιμές 37 δηλαδή δις σε τιμές φετινές και για την περίοδο 2021 μέχρι 2027. Να σας πω ότι με χαρά μου διαπιστώνω ότι είναι μεγάλη δέσμευση και κινούμαστε προς τη ζωστή κατεύθυνση. Σε τέτοιο επίπεδο όμως, επίπεδο φιλοδοξίας, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες για τα μεγάλα έργα υποδομών τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη βρίσκονται στη φάση του προγραμματισμού. Το Connecting Europe Facility επικεντρώνεται σε προγράμματα μεγάλης προστιθέμενης αξίας που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και ευρωπαϊκές υπηρεσίες και ευρωπαϊκά συστήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσει η χρηματοδότηση προφανώς και μετά το 2020 προκειμένου να είμαι και σαφής και να μην μακρηγορήσω να επικεντρωθώ στον κλάδο των μεταφορών του ΣΥΕΦ. Ένα από τους κλάδους λοιπόν ε, με μεγάλη προστιθέμενη αξία είναι ο συντηρόδρομο της Βαλτική, ε, μιας και είμαι ε, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη περαιτέρω Ευρωπαϊκή ενοποίησης σε ό,τι αφορά και τον τερματισμό των, της παράδοσης αυτής των παλαιών τρένων που είναι και αργά. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα που θα συνδέει την Φιλανδία με τις Βαλτικές, με την Πολωνία, ενδεχομένω και με τη Γερμανία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοινό τέτοιο πρόγραμμα στην ιστορία των χωρών της Βαλτικής. Μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να χρηματοδοτήσουμε ένα τέτοιο μεγάλο έργο και χαίρομαι που διαπιστώνουμε ότι το Rail Baltic είναι μία από τις προτεραιότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θα καλύψει ένας από τους τελευταίους ε, κρίκους που λείπουν ακόμα. Και πέρσι ο Επιτροπός Οτίνγκερ ανέφερε και το, ε, ε, το Rail Baltic και ένα άλλο πρόγραμμα και τόνισε ότι αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχα κονδύλια και τα δύο προγράμματα αυτά υπάγονται στο TNT, στα ευρωπαϊκά δίκτυα και για να μέχρι το 2030 θέλουμε να ολοκληρώσουμε τα προγράμματα TNT και αυτό θα δημιουργήσει 7,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης μεταξύ μέχρι το 2030 και 1,6% παραπάνω ΑΕΠ μέχρι το 2030. Είναι σημαντικό το ποσοστό αυτό. Αυτά τα έργα, ξέρετε, ποτέ δεν ωφελούν ένα, δύο, τρία μόνο κράτη-μέλη. Είναι κοινά έργα που ωφελούν όλους. Και αναμένεται στη Βαλτική να ολοκληρωθούν τα έργα μέχρι το 2024 μεταξύ Τάλιν, Ρήγας και Κάνας. Αναμένουμε να καταστεί λειτουργική γραμμή μέχρι το 2020 και μέχρι στη Βαρσοβία ε, το τελευταίο κομμάτι μέχρι το 2030. Για το λόγο λοιπόν αυτό, ο τομέα ε, των συνδροδρόμων θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη προτεραιότητα στο επόμενο ποδοπού και να υπάρχει και ιδιαίτερη χρηματοδότηση από το Connecting Europe Facility. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τις, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, γιατί είναι φιλικό προς το περιβάλλον, το μέσο αυτό μεταφοράς είναι ασφαλής με τρόπος μεταφοράς επίσης και έτσι συμβάλλει και στην ε, μείωση κατανάλωσης ενέργειας και στους περιβαλλοντικούς στόχους. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στις ε, τροπολογίες που θα καταθέσετε και σε μια επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ένας Ένα σκιώδη βλέπω μόνο για το θέμα αυτό. Ο κύριος Τόρβαλτς από την Άλτα. Έχετε δίκιο, πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να σας πω, ούτε και στους συναδέλφους έχω να πω πολλά για το θέμα αυτό. Προφανώς και ευχαριστούμε την εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της ε, προς τα θέματα που αντιμετωπίζουν ε, οι χώρες της Βαλτικής, τα οποία εν μέρη αγγίζουν και τη Φιλανδία. εμάς μας απασχολεί πιο πολύ το θέμα της διευκόλυνσης γιατί είναι συνδέοντα στην Ευρώπη. Και αυτό αποτελεί ένα γενικό στόχο εγκάρσιο που καλύπτει όλους τους ε, φακέλους. Θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Και πάλι θα σας απαντήσω στα σου ειδικά. Δεν βλέπω τέλεια και βλέπω ότι έκανα λάθος και οι σοσιαλιστές έχουν εδώ το σκιώδο τους. Ο κ. Πόπα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι καινούριο. Και καταλαβαίνω ότι ενδεχομένω να μην προσέξετε. Και όντω πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική γνωμοδότηση. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε επί της αρχής. Και οι τρεις πτυχές που αναφέρονται στην γνωμοδότηση θεωρώ ότι έχουν μεγάλη σημασία. Η συγγετρία έχει καταθέσει τροπολογίε και θα πρέπει να συζητήσουμε και τα αντίστοιχα ποσά για να δούμε τι αποφάσεις θα πρέπει να λεφτούν. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο ωστόσο και μπορούμε να οργανώσουμε τις συζητήσει μα με σωστό τρόπο. Θα συζητήσουμε λοιπόν κάποιες συγκεκριμένες πτυχές από κοινού και θα αποφασίσουμε προς τα ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Και η γραμματεία επίσης να πούμε ότι έκανε εξαιρετική δουλειά. Ε, Όπω και η συγκεκριά. Για την Κούα. Δεν ξέρω αν είσαστε σκιώδη, αλλά έχετε το λόγο. Ναι, βεβαίω είμαι σκιώδη τη ομάδα μου. Ο στόχο ε, σύνδεση τη Ευρώπη, ο εξευρωπαϊσμό των ε, μεταφορών και της ενέργειας ε, προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία εφόσον γίνεται με βιώσιμους στόχους και στόχους ε, γενικού συμφέροντος. Πρέπει να το διασφαλίσουμε αυτό. Ερώτηση. Εμείς θα υποβάλουμε μόνο τεχνικές τροπολογίες. Για παράδειγμα να μην γίνουν λάθη μεταξύ τρεχουσών τιμών και τιμών 18 ή θα υποβάλουμε και ευρύτερες τροπολογίες για τον έλεγχο της, ε, των βοηθειών που δίδονται για την, ε, τις μεταφορές ε, στο στρατιωτικό τομέα. Μήπως αν κάνουμε κάτι τέτοιο θα αφαιρέσουμε πόρους από τη σύγκληση. Αν ε, τώρα δω τα ενεργειακά θέματα, δεν θα πρέπει να δημιουργούμε υποδομές που δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικές. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών πρέπει να λαμβάνει και αυτά τα θέματα υπόψη της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τάραντ για τους πράσινου. Ευχαριστώ με την προσέγγιση, ε, συμφωνώ με την προσέγγιση της κυρίας Βάιντερε. Το μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη είναι σημαντικό πολιτικό μέσο της Ένωσης. Στηρίζω την προσέγγιση της, αλλά έχω δύο παρατηρήσεις. που είναι θέματα κυρίως της ε, Επιτροπής Μεταφορών. Στη χώρα μου, το 55% του πληθυσμού με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι κατά της ε, αδιαφανούς προώθησης ε, του Rail Baltica. Και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, γιατί τα άτομα που έλαβαν αυτές τις αποφάσεις ε, είναι δύο Εσθονοί. Η Εσθονή Επίτροπος και ένας Εσθονός που είναι μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Είναι παράδειγμα αυτό. Είπατε ότι θα δημιουργήσει 7,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Αυτό είπατε. Έχουμε 3 εκατομμύρια Λιθουανούς, 2 εκατομμύρια Λετονούς και 1 εκατομμύριο Εστονούς. Τι όλοι θα δουλεύουν στο σιδηρόδρομο. Άρα δεν θα μπορεί να έρθει κανείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ως Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ κύριε Τάραντ, λέει ο πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλο στο λόγο. Όχι. Λοιπόν. Λοιπόν. Χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι και ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολισμών θα γίνει στι 8 ή 9 Οκτωβρίου. Και η ψηφοφορία στην Ήτρε, η τελική ψηφοφορία, θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου. Οπότε κλείσαμε και το 4. Α, βεβαίως, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Αλλά και η Επιτροπή, αν θέλει. Ναι, ναι, σύντομα, λέει η συγγήτρια. Ευχαριστώ, Ίντρα. Είπα ε, θέση εργασία ερενούσα. Έτη απασχόληση. Εντάξει, ε, περιμένω τι τροπολογίες σας και για το συνάδελφο της ΓΚΟΕ. Βεβαίω έχουμε κάθε δικαίωμα να κάνουμε ό,τι τροπολογίες θέλουμε. Αλλά το κύριο είναι να συσπηρώσουν πλειοψηφία για την έκθεσή μας. Για την γνωμοδότησή μας δηλαδή. Παρακαλώ, κάντε τι τροπολογίε σα και ελπίζω ότι θα τι συζητήσουμε και θα καταλήξουμε και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Βάιντερ. Ωραία. Λοιπόν, τώρα περνάμε όντω στο 5. Το πρόγραμμα για το διάστημα και ο οργανισμός για το διάστημα της Ένωσης. Χάουερθ ο εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η πολιτική του διαστήματος είναι εξαιρετική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αξία περίπου 53 δις ετησίως. Απασχολεί 231.000 ε, ε, επιστήμονες ψηλών δεξιοτήτων και στον τομέα των ε, κατασκευαστικό της παραγωγής μάλλον. η τεχνική μας, τεχνολογική μας ανεξαρτησία και η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης είναι σημαντική για να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιες προκλήσεις όπως οι κλιματικές αλλαγές και να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε οικονομικό κέρδος προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Είναι Σημαντικό αυτό γιατί στον τομέα του διαστήματο τα προγράμματα είναι προγράμματα εταιρική σχέση δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και είναι και υψηλού κόστου. Οπότε χρειάζονται οικονομίες κλίμακας χάρη στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και προστιθέμενη αξία από την κοινή δράση των κρατών μελών. Επίσης, είναι επιτυχημένες οι προσπάθειές μας. Οι προσπάθειές μας ως τώρα με τον Γαλιλαίος, ε, το Γαλιλαίο και το Έγνος έχουν δώσει καλά αποτελέσματα στην ανεξάρτητη πλέγηση στο διάστημα ή για την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το πρόγραμμα παρατήρησης του Διεθνού Κοπέρνικος Αυτά που αντλούμε για την παρατήρηση των κλιματικών αλλαγών, την πολιτική αλλία, την επίτευξη των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη, όλα αυτά εξυπηρετούνται από τον Κοπέρνικο. Επίση, στην έκθεσή μου επικεντρώνομαι και σε δημοσιονομικά ζητήματα, διότι προφανώ αυτό είναι ο βασικό ρόλο τη Επιτροπή μα, να σχολιάσει τον προπολογισμό αυτών των προγραμμάτων. Απλώ ακολούθησα μια ε, προσέγγιση κάπως πιο ανοιχτόμυαλη από ό,τι κάποιοι θα υπέθεταν και θα σας πω γιατί. Πρώτον, διότι προσπαθούμε να είμαστε ε, σε μία βάση συνεπή με τους αριθμούς που προτείνουμε. Το 2018 οι προτάσεις που, κάνουμε, ε, που κάναμε ήταν σε τιμές Εκεί που υπάρχει κίνδυνος ως προς τον προπολογισμό είναι ίσως η δημιουργία ενός νέου κανόνα για τον οργανισμό που μέχρι τώρα το περισσότερο με, την, με τον εντοπισμό της γεωγραφικής και την, τον δορυφορικό συντονισμό. Γι' αυτό είχαμε αυτόν τον οργανισμό για τα διαστημικά προγράμματα τη Ένωση. Ω προ την υλοποίηση και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων, αυτά τα έβλεπε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός του Διαστήματος, που είναι εθνικός οργανισμός πέραν του πεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ μπορεί να υπάρξει κάποια επικάλυψη. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει κατά πόσον μπορεί να αξιολογήσει την ε, παραγωγή των ε, προγραμμάτων του διαστήματος, διότι όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνουν περιθώριο να παρέμβει κανείς στη δουλειά αυτή. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε και τη διπλή ε, δουλειά από διαφορετικούς οργανισμούς και τον διοικητικό συντονισμό ώστε οι δύο οργανισμοί να συντονίζονται και να μην ανταγωνίζονται. Εδώ είναι βέβαια θέμα και διατύπωσης, διότι η νομοθετική πρόταση είναι πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες και το πώς θα παρασκευάζονται ε, οι τεχνολογικές μας λύσεις. Βεβαίως, εδώ παίρνουμε και κάνουμε copy-paste από ανάλογες προτάσεις με σχετικές διατάξεις. Όμω, ε, η ιδιαιτερότητα του διαστήματο και των διαστημικών πολιτικών και των τεχνολογικών μέσων του είναι ότι συνήθω υπάρχει ίσω και μία μόνη πηγή ενό συγκεκριμένου τεχνικού μέσου σε ολοκληρό τον πλανήτη. Μπορεί να χρειαστεί να εισάγουμε από την Ελβετία, από τη ΣΥΠΑ, για κάποια ατομικά ρολόγια ή για κάποια ανταλλακτικά ή τέλο πάντων εξαρτήματα των δορυφόρων. Πρέπει να είμαστε πολύ ακριβεί ε, και στου όρου των δημόσιων προμηθειών, διότι δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε τα προγράμματα ή να πρέπει να βρούμε τρόπο να παρακάμψουμε τους κανονισμούς για να πάρουμε το εξάρτημα που μας χρειάζεται. Μας φαίνεται περιττό και γελίο κάτι τέτοιο γιατί θα ήταν και αρκετά διαφανές. Θα υποβάλω σχετικά τροπολογίες για το σχετικό δημοσιονομικό χαρτοφυλάκιο. Ε, επιζήτησα να μην αυξηθεί το ποσό πάνω από τις προτάσεις όσων ορίστηκαν στο πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα στοιχείο του προγραμματό που καλύπτει το ΣΑΤΚΟ και τα διαστημικά απόβλητα. Δεν είναι ένα θέμα που μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Αν δεν κανεί τι λεπτομέρειε, είναι μάλιστα αρκετά σοβαρό. Και ίσω και η αρμόδια επιτροπή να μπορούσε να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο για 500 εκατομμύρια σε όλη τη διάρκεια του πολιτού δημοσιονομικού. Ε, ίσως να μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό σε κάποια στιγμή. Και τέλος, για τον οργανισμό θα φροντίσω να το θέσω και στην ε, προσοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, αλλά το κοπέρνικος υποχρηματοδοτείται. Έχει πολύ λιγότερα από όσα χρειάζεται. Κάτι πρέπει να δούμε και να γίνει και γι' αυτό στο τέλο του ερχόμενου πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου. Σα ευχαριστώ. Και πάρε και το ροβάτι νοματικό σκιώδη ε, που έχει ζητήσει το λόγο. Θα ειδικά θα μιλήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα αφού το έχετε ρωτήσει τόσες φορές, φορές θα μιλήσω μας ικανοποιεί ιδιαίτερα η έκθεση την οποία μας παρουσίασε ο Τζον Χάουερθ. Συνήθως η συζήτηση για το πρόγραμμα το διαστημικό συγκεντρώνει τόση κριτική με την οποία όμως δεν συμφωνούμε γιατί πιστεύουμε ότι με τα διαστημικά προγράμματα μπορούμε να πετύχουμε μεγάλη εξοικονόμηση σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, θέματα γεωργίας, σε ό,τι αφορά την καταμέτρηση διοξυδίου του άνθρακα. Υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι να συνεχίσουν τα προγράμματα αυτά και θα υποστηρίξουμε. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε. Έχουμε λοιπόν δύο ερωτήσεις. Δύο θέματα μάλλον πραγματεύεται η έκθεση Χαουάρθα. Καταρχάς, όπως είπατε, οι τρίτες χώρες, την τροπολογία 12 είναι σημαντικό ο κίνδυνος η Ευρωπαϊκή, το Ηνωμένο Βασίλειο, συγγνώμη, να αποτελέσει τρίτη χώρα στο μέλλον. Και σε θέματα διαστημικών προγραμμάτων, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δραματίσει πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Θα πρέπει να επανέλθουμε, θεωρώ, στο θέμα αυτό ενδεχομένω και ύστερα στην τροπολογία 14. Ο εισηγητή προτείνει να υπάρχει μέλος ε, στην ε, ομάδα διαχείρισης. Είχαμε προβλήματα στο παρελθόν με το θέμα αυτό, αλλά θα δούμε κατά πόσον ε, από την άλλη δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τον κύριο Χάουαρτ. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να χαρήκατε που ακούσατε τα φιλανδικά σου ειδικά μου. Μάλιστα, υπάρχει μια εταιρική σύγχυση για το ποιος είναι ο σκιώδης από την κάθε πολιτική ομάδα παρά το γεγονός ότι ε, το σκέφτηκα ιδιαίτερα την προηγούμενη εβδομάδα και θεωρώ ότι ενδεχομένω ε, να μην πρόσεξα αρκετά γιατί το ΕΛΚΑ έχει σκιώδη και είναι η κυρία Χολμάιρη η οποία έχει και το λόγο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα βελτιώσουμε τις ε, επικοινωνίες μεταξύ του ΕΛΚ και της γραμματείας της Επιτροπής. Το ξέρει Τζον και αυτό αρκεί. Σας ευχαριστώ. Ο Τζον το ξέρει μάλλον. Ε, ευχαριστούμε, Τζον, που μας παρουσίασες και την γνωμοδότηση αυτή. Συμφωνώ απόλυτα. Για όλα, με όλα τα στοιχεία τα οποία ανέφερε. Και θα συνεχίσω το γερμανικά. Έχεις απόλυτο δίκιο που λες ότι ο Κοπέρνικος έχει έλλειψη χρηματοδότησης. Και θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο πιο λεπτομερώς τι γίνεται. Γιατί όταν ξεκινάμε με έλλειπη κονδύλια, τα πράγματα είναι μάλλον άσχημα. Δεν είναι σε δραματική κατάσταση, αλλά πότε θα αλλάξει αυτό. Αν το ξέρουμε και εφόσον το ξέρουμε, θα πρέπει να το συζητήσουμε για το πώς θα το επιλύσουμε το θέμα αυτό. Και τη χρηματοδότηση του Γαλιλαίου θα ήθελα να την εξετάσουμε και σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση σε κάποια χρονική στιγμή των δορυφόρων. Επίσης αυτό που λείπει, το έδειξες, είναι το θέμα της ΕΖΑ σε συνδυασμό με τα προγράμματα των υπηρεσιών τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι εδώ δεν θεωρώ ότι αντίκρινται να δημιουργήσουμε ανταγωνισμό. Νομίζω ότι πιο πολύ ενδείκνεται συντονισμό. Και αυτό ο συντονισμό θα πρέπει να υπάρχει εδώ και καιρό. Μία λοιπόν κοινή δομή συνεργασια από πλευρά τη ευρωπαικη Επιτροπής. Και γίνεται μία απόπειρα γενικά να ε, γίνει διπλή δουλειά σε ό,τι αφορά τα, τις αρμοδιότητες της ΕΖΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Να προσέξουμε, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να υπάρχουν συνέργειες, όσο πιο πολλές συνέργειες γίνονται μεταξύ των δύο τομέων. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, αλλά παρατηρώ ότι ο συντονισμός και η επικοινωνία μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν. να προσέξουμε να μην ε, πάνε σε άλλε υπηρεσίε, για παράδειγμα, διάφορε αρμοδιότητε και διάφορα καθήκοντα, τα οποία έω τώρα ήταν σαφώ ε, καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματο. Είναι καλό ο οργανισμό. Έχει αποδείξει την αξία του και, και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνεί, συμμετέχει. για τη τελική ανάλυση πρόκειται για έναν ε, διακυβερνητικό οργανισμό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει εντολέ και αναθέτει έργα στην Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν παρόλα αυτά να μην υπάρχουν ε, δουλειέ που γίνονται δύο και τρει φορέ, να μην ε, ξεκινήσει τελικά ένα ανταγωνισμό μεταξύ των υπηρεσιών. Θεωρώ ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελείται ο στόχο μα. Ε, κάτι άλλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα διαστημικά απόβλητα, είναι μια σοβαρή η διάσταση αυτή. σε ό,τι αφορά λοιπόν τα δεστημικά αυτά απορρίμματα, σημαντικό ζήτημα και θα πρέπει να κοιτάξουμε ακριβώ τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τι αναλύσει. Είναι πραγματικά περίεργο να, να λαμβάνει κανείς πληροφορίε, πληροφορίες, εικόνε, εικόνες. Καταλαβαίνει κανεί, ότι μπορεί και το διάστημα τελικά να μην είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζουμε. Και ότι και εδώ υπάρχουν κίνδυνοι για μας. Είναι προφανές το πρόγραμμα θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί σωστά, θα πρέπει να φροντίσουμε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να είναι ανταγωνιστική σε σχέση και με τα αμερικάνικα, σε σχέση με τα ασιατικά προγράμματα. Αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί και στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ε, επιδότηση που γίνεται σε άλλες χώρες για πυραυλούς και ό,τι καθεξής. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να, να φροντίσουμε να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού που δεν θα υπονομεύουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία και που θα προωθούν αυτές τις τεχνολογίες κλειδί. Και πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον τομέα αυτό και ελπίζω και από το Μάρτιο του 2019 να συνεχίσει να αποτελεί εταίρο στο Ηνωμένο Βασίλειο για να βρούμε μαζί κοινέ λύσεις και στο μέλλον. Ένα τελευταίο στοιχείο σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες downstream όπως ονομάζονται. Εδώ πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω προσπάθειες και να δούμε μήπως η υπηρεσία της Πράγας, η οποία είναι πολύ καλή υπηρεσία, πολύ κανός οργανισμός, μήπως θα μπορούσε να λάβει και ε, δορυφορικές υπηρεσίες, γιατί δεν ε, μπορούν να εκτελέσουν όλα τους τα καθήκοντα ενδεχομένω μόνο από την υπηρεσία της πράγας. Μήπως χρειάζονται λοιπόν και δορυφορικές υπηρεσίες σε άλλα κράτη-μέλη προκειμένου από κοινού με τον οργανισμό στην Πράγα να αναλάβουν την, ε, τα καθήκοντα αυτά. Να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χολμάιο. Αλλά επειδή πραγματικά δεν θέλω να εξαιρέσω κανέναν, να αποκλείσω κανέναν. Αν κάποιο άλλο θέλει το λόγο επ' αυτού, η Επιτροπή θέλει να προσθέσει κάτι. Α, θέλει. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ένα συνάδελφο από την DG, την Γενική Διεύθυνση Grow, θέλει να κάνει κάποια σύντομα σχόλια. Ναι, καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την εργασία η έκθεση πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, επιβεβαιώνει τον προϋπολογισμό που προτείνει η Επιτροπή. Δύο θέλω να σχολιάσω, δύο θέματα. Γιατί ετέθη το θέμα της διακυβέρνησης. Πρώτα απ' όλα, η δυνατότητα να διευρυνθούν οι δραστηριότητες του οργανισμού είναι πολύ περιορισμένες και αναλυτικά αναφέρονται στο σχέδιο κανονισμού και δεύτερον, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προτείνεται, είναι αυτή που ήδη ισχύει. Η Επιτροπή δεν προτείνει καμία αλλαγή επί των θεμάτων αυτών και θεωρώ ότι είναι λογικό το νομοθετικό όργανο να... Ε, δεν θεωρώ μάλλον ότι έχει έννοια να, το νομοθετικό όργανο να έχει θέση σε ένα τόσο τεχνικό θέμα μέσω συμμετοχής του Συμβούλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Να δώσω και πάλι το λόγο ε, στον κύριο Χάουαρθ για να ολοκληρώσει η συζήτηση, να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ όλους τους πήραν το λόγο. Καταλαβαίνω τι λέτε κύριε εκπρόσωπε της Γενικής Διεύθυνσης GROW. Εγώ απλώς θεωρώ ότι δεν ε, καθορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες και μπορούν να βελτιωθούν. Και αυτό επιχειρούμε με το κείμενό μας. Ευχαριστώ κύριε τόρβαλτ που θέσατε το θέμα για την ε, γεωργική παραγωγικότητα. Επισκέφθηκα το καλοκαίρι κάποιες γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου αξιοποιούν το Γαλιλαίο για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους κατά, την, ε, κατά τη συγκομιδή για να κάνουν ακριβώς στοχευμένη, στοχευμένο θερισμό αυτό ε, δείχνει πολύ συγκεκριμένα πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το Γαλιλαίο. Ναι, ναι. Το έχω υπόψη μου ότι μπορεί να γίνει τρίτη χώρα το Ρωμανό Βασίλειο. Κάπου, κάπου το πήρα είδηση. Χαίρομαι από αυτά που ακούω από την Επιτροπή σας, αλλά δυστυχώς σε διάφορα άλλα σώματα έχει υπάρξει μια καμψία και έχει δημιουργηθεί μια ανόητη κατάσταση για τον Γαλιλαίο. Και ορισμένοι βεβαίως θα μπορούσαν να υποχωρήσουν, αλλά αυτό θα σήμαινε ότι θεωρούν ότι κάπως θα εξευτελιστούν. Αν παρακολουθείτε το Βρετανικό τύπο και δεν θα σας κατηγορούσα εάν δεν τον παρακολουθήσατε, Υπάρχει η πρόταση η Βρετανία να φτιάξει το δικό της Γαλιλαίο. Για γέλια είναι αυτά. Κάτι για τους οργανισμούς που ανέφερε και η κυρία Χολμάιερ. Δεν θα πρέπει εμέσως να διευρύνουν τις αρμοδιότητές τους. Είναι κάτι που αυτόματα το κάνουν οι γραφειοκρατίες. Θέλουν να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερα καθήκοντα. Πρέπει λοιπόν να το περιορίσουμε. Ναι, ναι, οι αριθμοί είναι πραγματικά τρομακτικοί. Αν δείτε πόσα διαστημικά απορρίμματα υπάρχουν. Θα πρέπει οπωσδήποτε το πρόγραμμα να ξεκινήσει σωστά. Κάποιο στην Ήτρε απλώς πρέπει να δώσει μια σωστή αιτιολόγηση του γιατί πρέπει να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα και όχι μόνο δύο γραμμές σε μια τροπολογία. Και βεβαίως και έχετε δίκιο για το downstream servicing και φυσικά θα συνεργαστώ με τους κοιόδης ε, για να έχουμε μια σωστή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για τροπολογίες 3η 18 Σεπτεμβρίου 12 ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολισμών είτε στις 8 9 Οκτωβρίου και στην Ήτρε 21 Νοεμβρίου. Επόμενο θέμα. Επειδή βλέπω ότι παίρνετε όλο και περισσότερο, ε, μιλάτε όλο και περισσότερο όσο προχωράει η συνεδρίαση, σας παρακαλώ να είστε πιο σύντομοι, αλλά καλά φυσικά μην ε, ε τρέχετε πάρα πολύ. Πρόταση για κανονισμό και πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για, να, ε, για το ορίζον 20 και για την εφαρμογή του εισηγητή ο κύριο Τόρβαλτ. Όπω είπατε πρόεδρε και ευχαριστώ, παρουσιάζω δύο θέματα. Τον κανονισμό και την απόφαση για τον ορίζοντα του 2020. Όπω ξέρετε, είναι προτεραιότητα τη Ένωση μα η έρευνα και η καινοτομία. και λέμε συχνά ότι θέλουμε να είμαστε στην αιχμή ενό σωρού ε, πραγμάτων, όπως και στην Επιτροπή μας. Εδώ μιλάμε για προγράμματα που πρέπει να στηρίξουμε και ε, δημοσιονομικά, γιατί μέχρι τώρα μας έχουν δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Το Horizon 2020 ήταν πολύ επιτυχές ως τώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να το οδηγήσει σε μία ε, μετάλλαξη και μεταλλαγή όχι σε ε, επανάσταση. Οι στόχοι που έχουν ε, συμφωνήσει για τα κονδύλια και κρατών και κυβερνήσεων είναι ήδη μια αρχή, αλλά χρειάζονται περισσότερα. Και βλέπουμε και την ανησυχητική τάση μεταξύ των κρατών μελών να ε, υπάρχουν περικοπές της επενδύσεις για την καινοτομία και την έρευνα. Ιδίως όσο πιο πάνω πάει κανείς. Πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από αυτό το κακό συνήθειο. Τα δύο σχέδια γνωμοδότηση θα βρείτε την πρότασή μου να αυξηθεί το συνολικό ποσό του Horizon σε 120 δι σε σταθερέ τιμέ για το 2018 και νομίζω ότι είναι ένα ποσό το οποίο πρέπει να το προσπιστούμε. Κάποιοι θέλουν να πάμε ακόμη πιο ψηλά. Εδώ είναι από τα λίγα ποσά που ήμασταν τόσο ακριβείς ε, στην έκθεσή μας για τα επόμενα για τα υπόλοιπα ποσά του κανονισμού, μπορούμε να κοιτάξουμε την προσαρμογή του στον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή προτείνει συνολική ευελιξία 50% ε, για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμω το Horizon θέλουν ε, για κάποιο περίεργο λόγο να ε, περιορίσουν την ευελιξία σε 10%. Δεν καταλαβαίνουμε εδώ γιατί. Θα θέλαμε αυτό να προσαρμοστεί ώστε το πρόγραμμα να μπορεί να αυξηθεί κατά 15% αλλά να ε, υπάρξει περιορισμένη μείωση του 5%. Αυτό συνάδει με τις προτεραιότητες του προγράμματος για την Ένωση και θα το προστάτευε από ατυχήματα όπως οι περικοπές εξαιτία του ΕΦΣΥ. Όπως είπα και προηγουμένως, στη συζήτηση για το ΣΕΦ θα πρέπει να δούμε το 30% που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο ξανά και εδώ. Και στην απόφαση προτείνω να αλλάξουμε το πώς ε, είναι διαρθρωμένο το πρόγραμμα. Η αρχική πρόταση ε, είναι να υπάρχουν εφαρμοστικές πράξεις, επειδή όμως το πρόγραμμα περιλαμβάνει κανόνες για σημαντικά ζητήματα με σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις, τότε αυτό σημαίνει ότι οι κατεξουσιοδότητες οι πράξη είναι καλύτερες για την προσαρμογή των αρχών που ασχολούνται με την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Ε, είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω σχόλια και παρατηρήσεις για το πρόγραμμα της καινοτομίας και της έρευνας στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Τοιτς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να συγχαρώ τον εισηγητή που υποβάλει αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης, πρώτα απ' όλα για τις δημοσιονομικές πτυχές. Το χαρτοφυλάκιο του ορίζοντας 2020 είναι 91,4 δις ευρώ για το επόμενο, 94,1 ε, δις ευρώ για το επόμενο ποδοπού. Ε, το Κοινοβούλιο ήθελε να υπάρξει σοβαρή αύξηση. Εάν υπολογίσουμε τι θα συμβεί και το Brexit και η Μεγάλη Βρετανία και οι Βρετανοί ερευνητέ στα Βρετανικά πανεπιστήμια είναι βασικοί δικαιούχοι του Horizon 2020, τότε το ποσό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, το ερχόμενο, για την ερχόμενη επταετία, για το Horizon Ευρώπη 2007, με 27 ε, κράτη-μέλη, παρουσιάζει 50% αύξηση. Μάλλον 15% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο, την προηγούμενη φάση του Horizon 2020. Πρέπει να πούμε ότι βάσει του Horizon ε, και του ερευνητικού του προγράμματο δεν υπήρχαν ε, προγράμματα για ερευνητέ τη υπόλοιπη Ευρώπη. Επειδή λοιπόν έρχομαι από, από χώρα τη συνοχή, να ε, τονίσω ότι οι ερευνητέ από τα νέα εντό εισαγωγικών κατημέλη δεν παίρνουν μέρο σε τέτοια επιχειρημένα προγράμματα όπω το Horizon 2020. Θέλουμε αυξημένε, εντατικότερε προσπάθειε για να ενισχυθεί η συνεργασία των ερευνητών από χώρε με χαμηλότερε επιδόσει στην έρευνα και καινοτομία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γενογραφικέ τι γεωγραφικέ ανισότητε, την πρόσβαση των καταμελών στη χρηματοδότηση και να σκεφτούμε μια πρόταση για να βελτιωθούν οι χαμηλέ επιδόσει βάσει του Horizon 2020 και να καλλιεργήσουμε νέα κέντρα αριστεία. Τρίτον, ένα από τα βασικά στοιχεία του επτάετους κύκλου που θα ξεκινήσει το 2021 θα είναι η καινοτομία η καινοτομία που μπορεί να μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό κόσμο. Θα πρέπει να δώσουμε νέα, νέο βάρος στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων ε, και γνώσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία του αύριο για να αντιμετωπίσουμε περισσότερες προκλήσεις και να μπορούμε να ε, αποκομίσουμε ωφέλη από τις ερευνές της Ευρώπης για όλα τα κάτι μέλη. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Deutsch για την Σοσιαλιστές και Ο κύριος Χάουαρτ έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ και καλώς ορίζω την έκθεση του κύριου Τουρβάλ σε μεγάλο βαθμό. Θα συνεργαστώ με χαρά μαζί του για να καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση. Θα ξέρετε ότι είμαι υπέρ τη ε, διευρυνση του προγράμματος αυτού. Και θέλω αυτό να αποτυπώνεται στη γνωμοδότηση καθώς και την του Κοινοβουλίου για το πώς θέλουμε να διαμορφωθεί περαιτέρω και να διευρυνθεί ε, το πρόγραμμα αυτό, ορίζοντας ε, αποτυπώνεται και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, στα στοιχεία τα οποία μας παρουσιάστηκαν στο τέλος της διαδικασίας. Να αναφέρω επιγραμματικά κάποια, σημεία τώρα. Ο κύριος Τοίτσα έθεσε την αρχή, έθεσε μάλλον το θέμα α, της ε, συνέπειας του Brexit. Δεν θέλω να το συζητάμε συνέχεια για το θέμα αυτό, αλλά προφανώς για το πρόγραμμα αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, γιατί θα είναι σημαντικός ο αντικτύπος και ο αντίκτυπο τη ε, συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ελπίζω φυσικά να μην φύγουμε, αλλά η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου ως ε, τρίτη χώρα όπου θα συμβάλλει στο πρόγραμμα επί διαφορετικής βάσεως ε, σε σχέση με τη σημερινή αυτό θα ωφελήσει σημαντικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα το ίδιο. Ωστόσο, αν περιορίσουμε υπερβολικά τα κριτήρια βάσει των οποίων τα θεσμικά αυτά όργανα και να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι τα ερευνητικά κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι από τα κορυφαία του πλανήτη και είναι προς το συμφέρον όλων των υπόλοιπων ερευνητικών κέντρων που συνεργάζονται στα προγράμματα αυτά. Ουσιαστικά δύο πράγματα θα συμβούν. Θα μειωθεί η αξία του προγράμματος στο σύνολό του, θα περιοριστεί το επίπεδο αριστεία στα προγράμματα, το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί κριτήριο για το πρόγραμμα και θα μειωθούν και τα γενικότερα οικονομικά ωφέλη. Αν είμαστε, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ περιοριστικοί, θα ήταν λανθασμένη αυτή η προσέγγιση, θα πρέπει να την αποφύγουμε. Πάση θυσία. Επίσης, ε, να εξασφαλίσουμε ότι το επίπεδο των ε, συνεισφορών από τρίτε χώρε προς το πρόγραμμα θα αναφέρεται τακτικά στις αρχές της δημοσιονομικές ιδάλως, ενδεχομένω στο μέλλον να μην λαμβάνονται ενημερημένες αποφάσει για, το, για την πορεία του προγράμματος. Ελπίζω επίσης να προστατευτεί η έννοια α, του, της επιστήμης από μοτίμους μέσω ομοτήμων. Γιατί είναι ένα θέμα αυτό το οποίο προκύπτει στα συμβούλια. Χωρίς το στοιχείο αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει η επιστήμη. Και προσβλέπω στην εξέταση και των τεχνικών τροπολογιών του κ. Τορβάλτσα. Ένα τελευταίο σημείο. Κατανοώ γιατί χρησιμοποιείτε ποσοστιαίες μονάδες σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι ο κοινό θνητός δεν καταλαβαίνει τα ποσοστία, τις ποσοστίες μονάδες, τα στοιχεία για να καταλάβει. Και θεωρώ ότι ενδεχομένω αυτό να κάνει την έκθεση κάπω λιγότερο προσβάσιμη και θα ήθελα να το αποφύγουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Άλλο κανεί. Δεν έχουμε και χρόνο. Η Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Πολύ, πολύ σύντομα, αν θέλετε. Θα είμαι σύντομο, ε, πρόεδρε να επανέλθω στο θέμα του 10 και 15%. Να διευκρινίσω ότι το 10% που προτείνεται στην νομική βάση έχει να κάνει με την απόκληση την οποία μπορεί να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο. Ενώ το 15% είναι η διαθεσμική συμφωνία και άρα αποτελεί μια γενικότερη παρέκκληση η οποία δίδεται στην διάρκεια του προγράμματος στην αρχή δημοσιονομική. Είναι δύο διαφορετικά θέματα, λοιπόν. Να συμφωνήσω με τον κύριο Χάουαρθ ότι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτιμούσαμε να παραμείνουν τα ποσά αναπρόγραμμα και όχι οι ποσοστίες μονάδες. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο εύκολο και ευνοεί την κατανόηση. Ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος για την ε, ανακεφαλαίωση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή αλλά έχετε λίγο παραπάνω χρόνο μιας και λείπει η κυρία Χολμαϊέρ. Ευχαριστώ. Προς τον κύριο Ντόιτσε. Το έχουμε σκεφτεί το θέμα αυτό. Αλλά ένα τμήμα της Ευρώπης ε, προοδεύει ταχύτατα, ένα άλλο τμήμα όχι. Άμα δείτε για το, την έκθεση για τις βραδιπορούσες περι, περιφέρειες, θα δείτε ότι είναι πολύ ανησυχητικά τα στοιχεία για κάποιες περιφέρειες. Αλλά δεν μπορούμε να το λύσουμε λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πλέον να μας απασχολεί η αριστεία. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Και το συζητάμε με την Επιτροπή Περιφερειών για να βρούμε άλλο τρόπο για να καλύψουν την καθυστέρηση κάποιοι βραδιπορούντες. Θα τα συζητήσουμε μαζί προσεχώς. Αναβερθήκατε στα θαυμάσια πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχει πρόβλημα εδώ τώρα για ποσοστά και ποσά. Για τεχνικό λόγο χρειαζόμαστε τα ποσοστά γιατί είναι ευκολότερο να μετατραπούν κατόπιν σε αριθμούς. Αλλά όσοι εμένουν στους αριθμούς, θα σας δώσουμε και τους αριθμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και πάλι το χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών 8 ή 9 Οκτωβρίου, στην Ήτρε 21 Νοεμβρίου. Κλείσαμε τα 6 και 7. Τέλος η πολιτική κτηρίων. Η κυρία Χόλμαρ δεν είναι εδώ. Και πρέπει να τελειώσουμε στις 11. Ναι, ήθελε να πει ότι θέλει μια παράταση. Να παραταθεί η προθεσμία για να ληφθεί απόφαση για την πρόταση για το JMO2 και τα Eurofis. Δύο εβδομάδες, κατά δύο εβδομάδες. Οπότε, ωραία, αναβάλλεται η λήψη απόφαση για δύο εβδομάδες. Αυτό ήθελε να μας πει. Ωραία. 9, 10 και 11 για ψηφοφορίες για διάφορα σημεία του προπολογισμού, αλλά επειδή δεν έχουμε αιτήματα μεταφορών για τα θέματα αυτά, μεταφορών πιστώσεων, λοιπόν τελειώνει η συνεδρίασή μας, πολύ ωραία, και μετά θα αναλάβει ο πρόεδρός μας, ο κύριος Αρτουή, για τη συνεδρίαση των συντονιστών, που έπεται αμέσως ευχαριστώ.